εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ο Φραντσέσκο Σιλβέστρης έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Στι τελευταίε εβδομάδε πολύ σοβαρές ε, βροχοπτώσει έχουν πλέξει διάφορες ε, ευρωπαϊκές χώρες και έχουν γονατίσει τους ε, εκεί πληθυσμού. Έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Βέλγοι στο, στο Μπραμπάντ και στην, στη Δυτική Φλάνδρα. Ήταν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δέκα ετών. Έπεσαν, υπήρξαν βροχοπτώσει τόσο σημαντικέ όσο καταγράφονται κατά τη διάρκεια τριών μηνών. Παρόμοια κατάσταση στη Γαλλία, όπου πολλές, ε, πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, έχει μπλοκαριστεί το σύστημα των μεταφορών, έχουν κλείσει διάφορες ε, σύραγγε λόγω ε, ακόμα και σιδηροδρομικέ γραμμέ. Πριν από 20 μέρες στην Ιταλία χτυπήθηκαν οι περιφέρειες της, του Βένετο με δύο νεκρού, η Λιγκούρια, η Καλάβρια, το Σαλέρνο, η Καμπάνια και η Τοσκάνη. Επίσης ε, ένα άτομο χάθηκε στο Ροβίγα. Εκατομμύρια ευρώ μόνο για τις άμεσες παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν, ε, ακόμα δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις για το ποιες, ε, ποιο είναι το κόστος των καταστροφών. Επίσης υπάρχουν 500 εξοπλισμένοι άνθρωποι τουλάχιστον. Υπήρξαν ζημιές όσον αφορά τα ζώα και τις καλλιέργειες. Πρέπει να κινητοποιηθεί η βοήθεια και η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη ήδη λειτουργήσε που ο κόσμος βοήθησε τους πληθυσμούς που επλήγησαν στις πρώτες κρίσιμες ε, στιγμές. Η δεύτερη πτυχή, η Πρόεδρε, συνδέεται με τις επιπτώσεις μακράς διαρκείας ε, αυτών των καταστροφών ο ευρωπαϊκός ε, Ιστό αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχασαν τα πάντα, δηλαδή μηχανήματα αλλά και πρώτε ύλε. Το ίδιο και με τους γεωργού που έχασαν τα τρακτέρ τους, τις μεταμηχανήματά τους, τους πόρους. Ε, επίσης ε, χάθηκαν χιλιάδες ζώα. Αυτές οι επιχειρήσεις που ήδη αγωνίζονταν με την οικονομική κρίση βρίσκονται πια στα πρόθυρα τη πτώχευση. πράγμα το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα έχει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα διαλύσει τον ε, ε, ιστό το βιομηχανικό της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, ακόμα και κατ' εξαίρεση ε, και ακόμα και αν δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2011 πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο δράμα και που έχουν το δικαίωμα να αισθανθούν την αλληλεγγύη αυτού εδώ του Κοινοβουλίου και την ευρωπαϊκή στήριξη. Τρέλα. Κυρία Εστρέλα, από τους ε, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών, εγώ θέλω να δηλώσω την αλληλεγγύη μας για όλες ε, τις περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και θέλω να, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Το 2010 μας βρίσκει μπροστά σε κατάσταση σοκ ενώπιον των της καταστροφής που συνέβη στην Μαδέρα. Αμέσω μετά ε, χτυπήθηκε η Γαλλία. Μετεωρολογικά ακραία φαινόμενα έχουν επίσης πλήξει την Ισπανία, την Βέλγιο, την Γερμανία, τις κατοχώρες και προκάλεσαν ε, τεράστιες ζημιές. Στην κεντρική Ευρώπη οι πλημμύρες του καλοκαιριού κάθε φορά είναι πιο συχνές και καταστροφικές. Στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και διάφορα εργοστάσια και βιομηχανίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Ε, στην ε, Νότια Ευρώπη κάθε χρόνο εκατοντάδες εκτάρια δάσους ε, αναλώνονται ε, από τη, από, τη φωτιέ, από τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Κάθε φορά βλέπουμε μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές με μεγαλύτερες σημειές σε ανθρώπινες ζωές, σε περιβαλλοντική επιδείνωση και οικονομική επίσης, οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να, να προλάβουμε, να, κάνουμε, να ασκήσουμε ε, προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και την αρμόδια υπηρεσία, η καλύτερη διατήρηση των οικοσυστημάτων και η καλύτερη διαχείριση των παρακτήων ζωνών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Εξάλλου, οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας θα πρέπει να ενισχυθούν και τα κοινοτικά μέσα ανταπόκρισης θα πρέπει να απλοποιηθούν και να ισχύσουν ε, πιο ευέλικτοι κανόνες ε, εκτέλεση και εφαρμογή του. Μιλάμε για το Ταμείο αλληλεγγύη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το Συμβούλιο εξακολουθεί να εμποδίζει το νέο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύη που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Να θυμίσω επίση ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την εξηρασία, για να μπορέσουμε να, να εκπαιδεύσουμε καλύτερα προσωπικό και να παρατηρούμε καλύτερα τα διάφορα φαινόμενα. Έτσι μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους ε, φιλελεύθερους, ο κύριος Ντέρκ Στέρξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε συλληπιτήρια στα θύματα. Στη χώρα μου πνίγηκαν τέσσερα άτομα και σε άλλες χώρες πλήγησαν χιλιάδες άνθρωποι, οπότε η σχέση μας γίνει πρώτα απ' όλα σε αυτούς. Τις ε, μέρες, ε, εβδομάδες και χρόνια πέρασαν υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα βεβαίως με πλημμύρες ε, και έχω ένα ερώτημα προς την Καμισιόν. Στην αξιολόγηση των τωρινών γεγονότων θεωρείται πως ε, θα είναι λογικό να έχουμε ειδικού από τα διάφορα κράτη-μέλη και της ε, περιφέρειας ε, και να ακούσουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για το τι συνέβη για να δούμε καλύτερα τα αίτια. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Εάν καταλάβουμε καλύτερα τα αίτια, νομίζω θα μπορέσουν έτσι να μιλήσουν και οι ειδικοί για μέτρα. Να γίνει μια ανάλυση κινδύνου ανά περιοχή και λεκάνη απορροής όπως κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προλάβουμε αυτές τις ε, καταστροφές. Και τέλος, όταν έχουμε ξανά μια τέτοια κατάσταση, να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα αυτά τα μέτρα. Οπότε νομίζω καλό θα είναι εδώ πέρα να ακούσουμε τους ειδικού για να αξιολογήσουμε το τι συνέβη αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρος, κυρία Ιζαμπέλ Ντουραν των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα εκ μέρους των Πρασίνων να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες, σε όλα τα άτομα τα οποία επλήγησαν από τις φοβερές αυτές πλημμύρες, όσους έχασαν ένα αγαπημένο πρόσωπο ή μέρος της περιουσίας τους. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσουμε όλους ε, τους διασώστες, τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που δραστηριοποιήθηκαν ε, σε όλες αυτές τις πληγήσεις περιοχές. Θα πρέπει όμως και στο μέλλον να βοηθήσουμε τους πληγέντες, του αποζημιώσουμε, αλλά να ε, υιοθετήσουμε και μια καινοτόμο τολμηρή πολιτική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματο. Προτείνω λοιπόν τρία είδη μέτρων στην Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, δημιουργία σχεδίων κατασκευή καινοτομία, τα οποία θα οδηγήσουν σε αδιαβροχοποίηση του εδάφου. Γιατί όταν δημιουργούμε ένα εμπορικό κέντρο, ένα νέο οικισμό κτλ., θα πρέπει να φροντίζουμε την αδιαβροχοποίηση του εδάφου λίγο περισσότερο. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για ε, τις ε, ζώνες που μπορούν να υποστούν πλημμύρες. Επίσης, γεωργική πολιτική, γιατί σίγουρα υπάρχει ε, ευαλωτότητα του εδάφου λόγω και των καιρικών συνθήκων. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα λοιπόν. Και τέλος, συναγερμός, συντονισμός των τοπικών αρχών για την πρόληψη ή αποτροπή αυτών των καταστάσεων. Νομίζω ότι πολλές φορές δεν υπάρχει επαρκώς ταχεία ενημέρωση, ούτε καλή, καλό συντονισμός έπρεπε λοιπόν και οι προειδοποιήσει τη Μετρολογικής υπηρεσία να διαδίδονται πολύ πιο γρήγορα. Πρέπει στο σύνολο των πολιτικών αυτών να υπάρχει το σκέλος και τη πρόληψη ε, και τη ενεργού πολιτική. Θα πρέπει επίση να δημιουργηθούν ε, και πιο χρήσιμε πολιτικέ διότι όταν θα έχουμε πάλι κάποιο ε, ακραίο μετρολογικό φαινόμενο θα είμαστε πάλι εδώ για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μα, επιχειρήσει οικογένειες και νομίζω ότι για να το αποφύγουμε αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία σε όλες μας τις πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκέρλινγκ, από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η ομάδα μου βεβαίως ε, συλληπείται τα θύματα. Έχω προσωπική εμπειρία. Υπήρχε μια πλημμύρα στην δική μου την περιοχή, η οποία πρώτα απ' όλα με έφερε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ενέπνευσε να γίνω βουλευτής. Οπότε η κινητοποίηση τότε του Ταμείου Αλληλεγγύης ήταν μεγάλο γεγονός για μένα. Και αυτή την εβδομάδα πάλι στην Κορνουάλη είχαμε πλημμύρες. Αυτό το οποίο ήθελα να πω το είπε ο κύριος Στέρξ, αλλά πρέπει να το επαναλάβω. Θεωρώ πως είναι σημαντική η έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά ξέρουμε πόσο γρήγορα αλλάζει και κινείται ο καιρός και αναρωτιέμαι αν είναι σωστή χρήση των κονδυλίων το να αφιερώσουμε πολλά λεφτά στην έγκυρη προειδοποίηση για τον καιρό που υπάρχει ήδη. Το θέμα είναι τι κάνουμε όταν έχουμε την προειδοποίηση. Και θεωρώ, όπως είπε και ο κύριος Στέρξ, πως μπορούμε να μάθουμε πολλά, οπωσδήποτε η Ευρώπη μπορεί να μάθει πολλά, και να υποφεληθεί με το να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Και ξέρω πως στην περίπτωση του sir από το οποίο κατάγομαι, Οφεληθήκαμε από τις επαφές μας με αυστριακές περιοχές που είχαν τεράστια εμπειρία σε πλημμύρες, σε υψόμετρο που εμείς δεν είχαμε. Καλή ιδέα λοιπόν θα ήταν η Κομισιόν να κάνει κάποιες περιφερειακές συνδέσεις για να διδαχτούμε ο ένας από τον άλλον γιατί σαφώς δεν θα εξαφανιστεί το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ για την Ενωμένη ΕΕ, Ευρωπαϊκή Αριστερά ο κ. κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Γκουε θα ήθελα και εγώ να συλληπιθώ τα θύματα. Συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα σε αυτό και συμφωνούμε επίσης στο ότι πρέπει να βοηθήσουμε γρήγορα. Και ακούσαμε αρκετά λογικά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβω αλλά τα υποστηρίζω. Μία πτυχή θα ήθελα να τονίσω, οι μακροπρόθεσμες ζημιές δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάποιες φυσικές επιπτώσεις είναι πιο μακροπρόθεσμες από όσο μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό μου φαίνεται σημαντικό να προσέξουμε για τη μακροπρόθεσμη αυτή καταστροφή της φύσης και της ε, φυσικές αυτές καταστροφές. Αλλά εδώ μπορούμε να συζητάμε, αλλά νομίζω το καλύτερο είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να βοηθήσουν τον εαυτό τους επιτόπου. Γιατί ξέρουν καλύτερα τις συνθήκες επιτόπου από ότι εμείς από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μάρα Μπιτσότο από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου εξ ονόματος της ομάδας μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρε. 5 εκατομμύρια κάτοικους έχει η δική μου περιφέρεια, όπου 500.000 επλήγησαν από τις πλημμύρες. 7.000 ε, έχουν εκτοπιστεί, έχουν ε, πλημμυρίσει εκατοντάδες ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πολύ σοβαρές ζημιές υπέστησαν οι επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι διαστάσεις αυτής της καταστροφής η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα. Πρέπει να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης και γνωρίζουμε ότι αν δεν εγκριθεί ο προπολογισμό, το Ταμείο αυτό δεν μπορεί να κινητοποιηθεί. Μα η Ευρώπη πρέπει πέρα από το να μιλάει εδώ για μεγάλες στρατηγικές, για προγράμματα ανάπτυξης και προγραμματισμούς ε, φαντάσματα, να επενδύσει περισσότερο στην ε, έρευνα, να ε, εκτιμήσει τους γεωλογικούς, υδρογεωλογικούς κινδύνους, να εγκαθιδρύσει ένα προληπτικό σύστημα άμυνα να δημιουργήσει όσον αφορά το νερό για να μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες. Ελπίζω πραγματικά πως η Ευρώπη για μια φορά θα δώσει μια απάντηση και θα ακουστεί περισσότερο και να μην μείνει απομακρυσμένη από τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Uh, uh, thank you. Thank Σας ευχαριστώ κυρία μου. Εδώ Ολοκληρώνεται η συζήτηση, η σύντομη αυτή συζήτηση για τις ε, πλημμύρες στην Ευρώπη φέτος.